Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω να ανακοινώσω μια τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση της Επιτροπής για τις μεταφορές αποβλήτων, δεν μπορέσαμε να το συζητήσουμε χθε το απόγευμα. Θα προσθεθεί σήμερα ως τελευταίο θέμα στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θα τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη με την τροποποίηση αυτή. Προχωράμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων. Ε, θα ψηφίσουμε πάνω στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μπριάνο. Θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω ότι έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία για τις τροπολογίες 13 και 72. Συμφωνείτε? Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ε, αν συμφωνείτε. Ποιος είναι υπέρ ε, της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ποιος είναι κατά. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας λοιπόν. Okay, the vote is Λήξη της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτό το αίτημα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα, θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, όχι, λάθος. Ένα λεπτό να εξηγήσω. Θα πρέπει να συμφωνήσουν 17 συνάδελφοι με το αίτημα. 21 συνάδελφοι υπερψήφισαν. Έτσι γίνεται δεκτό το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, περιοχή των Άλπαιων. Συμβαστική 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Τελευταίο τμήμα ως προσθήκη στην α, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση αν θέλετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 37. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία μάλλον συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 ηλεκτρονικά με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 77 υπέρ, κατά Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 77. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 89 και αυτή σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 99, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 104 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 104. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 105 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται.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 κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 12 πέρας απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 13 με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρακαλώ, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην ε, συναδελφό μας, την κυρία Μπριάνο. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να φτάσει ο Επίτροπος Άριας Κανιέτε. Αγαπητοί συναδελφοί, μπορούμε να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μιγγέλ Κανιέτε, ο οποίος είναι ο Επίτροπος για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Είναι τμήμα λοιπόν του διαρθρωμένου μας διαλόγου. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρα συζήτηση στα πλαίσια του ετήσιου διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Κομισιόν και της Επιτροπής ΕΝΔΙ. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2006 τα θέματα που μας ε, ενδιαφέρουν και φυσικά και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, μετά από τη συμφωνία που έγινε στο Παρίσι πέρσι, ο στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων να μάθουμε και για την πρόοδο στην προτινόμενη νομοθεσία για να προσαρμοστεί το πλαίσιο στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, η, ο επιμερισμός προσπάθειων, αντιμετω, αντιμετώπιση της αλλαγής χρήσης γης, γεωργία κτλ. Η Επιτροπή μας θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά την εφαρμογή των ε, στόχων του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και η πρόθεσή μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνεκτικότητα με τις υποχρεώσεις που συνήθισαν στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά για τις προκατακτικές σας παρατηρήσεις και θα αρχίσει φυσικά ο γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη. Είναι μεγάλη τιμή να έχω αυτή τη συζήτηση μαζί σας σε μια ιδιαίτερη στιγμή την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων στη Νέα Υόρκη. Για μένα είναι ακριβώς η στιγμή που τελειώνουν οι πανηγυρισμοί και ερχόμαστε στην εφαρμογή των αποφάσεων. Το 2016 θα είναι ένα σημαντικό έτος διότι προετοιμαζόμαστε <clears throat> για την εφαρμογή του πλαισίου για το 2030 και την επίτευξη των στόχων μας. Έχουμε κάνει ήδη τις πρώτες προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των υποχρέωσεων που έχουμε αναλάβει με την ε, δέσμευση συγκεκριμένη της τροποποίησης του συστήματος για την εμπορία κομμών. Ξέρω ότι ο κύριο Ντάνκαν και οι σκιώδεις εισηγητές επεξεργάζονται το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο βήμα είναι να αντιμετωπίσουμε τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ETS. Πώς θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε την αλλαγή της χρήσης γης, και την δασοκομεία. Όλα αυτά τα νέα στοιχεία θα παρουσιαστούν πριν από το καλοκαίρι μαζί με την πρότασή μας για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Και παράλληλα θα παρουσιάσουμε μια ανακοίνωση για την μείωση της χρήσης άνθρακος στις μεταφορές. Το 3ο 4 ο του 2016 η Κομισιόν θα το πακέτο για την ενεργειακή απόδοση που περιλαμβάνει και μια αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση με στόχο να επικαιροποιήσουμε την πολιτική μας στα θέματα της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας ώστε να αντανακλάται και ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030. Το τέταρτο τρίμηνο θα παρουσιάσει το νέο πακέτο για τα θέματα των ε, ανανεώσιμων ενεργειών και την πολιτική βιωσιμότητα και αηφορίας μετά το 2020. Θα εξεταστεί επίση και το θέμα ενό ισχυρού μηχανισμού διακυβέρνηση για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί που έχουν θεσπιστεί και αυτό περιλαμβάνει τους στόχου ενέργειας και κλίματος του 2030. Το 2016 λοιπόν εμείς θα πρέπει να έρθουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία για την διακυβέρνηση της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Και μετά από τη συνέλευση του ΙΚΑΟ το Σεπτέμβριο, η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια έκθεση και εάν υπάρχει ανάγκη προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από, την, από τον αεροπορικό κλάδο. Να πω τώρα σε πιο πολύ λεπτομέρεια για αυτές τις ε, προτάσεις. Καταρχήν οι προτάσεις για την αλλαγή γης και ο επιμερισμός προσπαθειών. Η Κομισιόν έχει συμφωνήσει ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό μείωσης κατά 40% των αερίων του θερμοκηπίου οι τομείς οι οποίοι βρίσκονται εκτός του ETS, μεταφορές, κτίρια και γεωργία, θα πρέπει να, έχουν, να υποστούν μείωση κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2005. Εφέτος θα υποβάλουμε μια πρόταση για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση σε εθνικούς στόχους και στη συνέχεια μετά από τις κατευθυντήρες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα καθοριστούν οι εθνικοί στόχοι επί τη βάση του ΑΕΠ κατά κεφαλήν και επιπλέον για τα κρατη που έχουν ΑΕΠ κατά κεφαλή πάνω από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσαρμοστούν οι στόχοι για να υπάρξει σωστή και δίκαια κατανομή επί τη βάση του ισχύες κόστους κόστους-οφέλους και της ε, σωστής κατανομής μεταξύ των μελών κρατών. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα, είναι, ε, θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα να υπάρξουν ε, μειώσεις οι οποίες να μην είναι πολυδάπανες για τα κάτι μελη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η γεωργία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%. Η σημασία της γεωργίας και του τομέα της αλλαγής χρήσης γης είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να παραμείνουμε κάτω από το στόχο του, των δύο βαθμών αύξησης θερμοκρασίας επί τη βάση του, των αποφάσεων του Παρισιού. Θα πρέπει λοιπόν Να, να ενσωματώσουμε και την αλλαγή χρήσης γης στις ε, ε, αλλαγές που θα εφαρμόζουν. Θέλουμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετριασμού στη γεωργία και την ανάγκη να λάβουμε υπόψη και τι εκπομπέ που προέρχονται από την αλλαγή τη χρήση γη. Μαζί με τον Επίτροπο Χόγκαν έχουμε έρθει σε διμερέ επίπεδο σε επαφή με 19 υπουργού. Το να ακούσουμε τι απόψει σα σήμερα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο τη προετοιμασία τη πρόταση τη Κομισιόν τον Ιούλιο. Εμεί βασιζόμαστε λοιπόν στο πλαίσιο του Λούλου δηλαδή για την αλλαγή τη χρήση γη και την ε, δασοκομεία, ώστε να έχουμε μια αξιοποιημένη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευκαμψία ενώ συγχρόνω διαφυλάσσει την ακαιρεότητα του περιβάλλοντος. Όλα τα κράτη-μέλη είναι φυσικά υπεύθυνα για να επιτύχουν τι μειώσει στους τομεί αυτού πέραν του συστήματο αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξουν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε σε όλου του τομεί τι μειώσει αυτέ η μείωση της Χρήση άνθρακος στη μεταφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε φιλόδοξου, συνεκτικούς και καινοτόμους στόχους και πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσουμε τη μείωση της χρήση άνθρακα στον τομέα μεταφορών. Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση θα πρέπει να υπάρξει δράση για αυτή τη μετάβαση. Σε επίπεδο εθνικών περιφερειακών και τοπικών αρχών και σε επίπεδο πολιτών, αλλά φυσικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την πρόταση αυτή για την, τον επιμερισμό των προσπαθειών, θα παρουσιάσουμε μια ανακοίνωση για την μείωση τη χρήση άνθρακο στι μεταφορέ, που θα αναφέρει πόσο το μέσο μεταφορών μπορεί να συμβάζει στην επιτεύξη των στόχων του 2030. Η ανακοίνωση αυτή καλύπτει όλου του τομεί μεταφορών. Για την μείωση λοιπόν της χρήσης άνθρακος, η ανακοίνωση θα τονίσει ιδιαίτερα τη μείωση τις περιεκτικότητας σαν τα στα καύσιμα και τα αναλλακτικά καύσιμα, την καλύτερη διαχείριση των ε, μορφών οδικών μεταφορών και την μετακύληση των ε, μεταφορών σε άλλες μορφές ε, μεταφορών και επίσης την δημιουργία πλαισίων και προδιαγραφών για τις δοκιμασίες οχημάτων και την αναθεώρηση του τωρινού κύκλου δοκιμασιών. Το να έχουμε φιλόδοξες, αξιόπιστες και ρεαλιστικές προδιαγραφές για τις εκπομπές επέκεινα του 2020 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 και να ε, οδηγήσουν καιρό στην επίδευξη των στόχων του 2050. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν και σε μία πρόταση για νέα ε, πρότυπα εκπομπών για τα αυτοκίνητα, ε, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και τα αυτοκίνητα μέχρι το 2017. Ο στόχος είναι να επιτύχουμε και στόχους οι οποίοι θα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την καιροτομία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. θέλω να υπογραμμίσω τις προσπάθειες που έχει κάνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία τα τελευταία χρόνια και την προσθέμενη αξία που έχει προσποριστεί με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή οικονομία. Ξέρω ότι περαιτέρω ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών στα αυτοκίνητα θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε, αλλά μπορούμε να πετύχουμε ρεαλιστικού και αξιόπιστους στόχου. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαδικασία δοκιμασία των οχημάτων σε σχέση με τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρωπου. Μετά από το σκάνδαλο τη Volkswagen είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη όλων σε ό,τι αφορά τι μετρήσει και τι δοκιμασίε για τι εκπομπέ. Γι' αυτό τώρα προχωρούμε στην εφαρμογή της εναρμονισμένης παγκόσμια διαδικασίας ελέγχου για τα ελαφρά οχήματα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν πιο ε, και πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες ε, ε, δοκιμασιών. Θα έχουμε με τον τρόπο αυτό πιο ρεαλιστικά και πιο αξιόπιστα στοιχεία και η Κομισιόν θεωρεί ότι μπορεί αυτή η νομοθεσία να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό. Και επίση η Κομισιόν θέλει να μειώσει και τι ε, πομπές από τα βαρέα οχήματα επεξεργαζόμαστε μια πρόταση για την παρακολούθηση και την, ε, τις ε, εκθέσεις που πρέπει να, να παρέχονται, η οποία πρέπει να εγκριθεί το 2017, ώστε να έχουμε περισσότερες γνώσεις για τις ε, εκπομπές των βαρέων οχημάτων σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακος. Και επίσης η Κομισιόν θα εξετάσει και τη δυνατότητα να αναπτύξει ειδικού στόχους για τα βαρέα οχήματα. Αξιότιμα μέλη λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως βλέπετε αυτή θα είναι μια πάρα πολύ έντονη χρονιά σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα θέματα Τη κλιματική αλλαγή, και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μετά από τη Συμφωνία των Παρισίων ή έχουμε κάνει μια πολύ καλή εκκίνηση και αν μπορέσει να εγκριθεί όλη αυτή η νομοθεσία θα είμαστε σε ένα σημείο καμπής για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα την συζήτηση από πλευρά των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Πίτερ Λίζε από το ΕΛΚΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εισαγωγή σας ε, και ε, για την ε, δουλειά που κάνετε. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Διεξάγεται έντονη συζήτηση τουλάχιστον εντός της πολιτικής μας ομάδας υπάρχει μία πρόταση από πλευράς ε, ε, της ε, βαριάς βιομηχανίας σχετικά με ένα 10% ε, συνολικά 43% μείωση. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε οι καλύτερες επιχειρήσεις ε, στις βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας όπως για παράδειγμα τη βιομηχανία του Χάλιβα. Αν ανήκουν ε, λοιπόν στο καλύτερο 10% ε, να ε, έχουν ε, αποζημίωση 100% όσον αφορά τις δαπάνες τους. Όσον αφορά τον επιμερισμό της προσπάθειας, τα κράτη-μέλη διστάζουν να αναλάβουν ευθύνη. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να είσαστε πολύ αυστηρός και να μην αφήσετε τα κράτη-μέλη ε, να ξεφύγουν. Δεν μπορεί κάποιοι τομείς ε, της βιομηχανίας να ε, επιβαρύνονται ενώ οι βιομηχανίες για τις οποίες είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη να περνούν πιο εύκολα. Και όσον αφορά την Λουλουσιέφ, τη χρήση γης και αλλαγή στη χρήση γης και δασοκομεία, να μην επιτρέψετε να υπάρξουν πολλά παραθυράκια. Και τέλος, ε, όσον αφορά τις αερομεταφορές, συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα εμπορία εκπομπών, ε, δεν καλύπτονται όμως με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και άλλοι τομεί. Είναι λιγότερο φιλόδοξοι η στόχοι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ήταν όμως χρήσιμο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να αντιμετωπίσουμε τις αερομεταφορές με τον ίδιο τρόπο ε, που αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ε, τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ματίας Χρότε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά την ωραία αίσθηση που είχαμε στο Παρίσι, όπου δεν υπολογίζαμε τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις ε, άλλωστε γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε σε πράξεις και να προωθήσουμε την ε, αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ο συνάδελφος ε, από το και ανέφερε του τομεί όπου θέλει να υπάρξουν ε, παρεκκλήσει, αλλά εγώ δεν θα ήθελα παρεκκλήσει ε, στι αερομεταφορέ. Είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ο καθένα πρέπει να πληρώνει για το αυτοκίνητό του, το βενζινάδικο θα πρέπει να πληρώνει, αλλά ειδικά οι αερομεταφορέ όπου δεν πληρώνονται φόροι και δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σχετικό μέσο να να παράσουμε μια παρέκκληση διότι θα ξεκινήσει η συζήτηση γιατί ε, να έχουν τέτοια προνόμια. Χρειαζόμαστε λοιπόν η μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το σύνολο του συστήματος εμπορίας εκπομπών και ιδιαίτερα τις αερομεταφορές. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στο Παρίσι ε, είχε πολύ σημαντική παρουσία. Δυστυχώ όμως αποδυναμώθηκαν τελικά τα επιχειρήματα όσον αφορά τα πρότυπα για το διοξίδιο του άνθρακα. Στις ε, μεταφορές στα βαρέα οχήματα και στα ελαφρά οχήματα, τα ιοταχή. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης ε, όσον αφορά τα τίζελοκίνητα αυτοκίνητα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ποια αυτοκίνητα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα πρέπει να γίνει κάτι στον τομέα αυτόν. Με την έγκριση τύπου δεν ε, θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα μόλις στο αέρα που έχουμε στη Βόρεια Ιταλία, που έχουμε ε, στις πόλεις, εάν υπάρχουν ε, παραθυράκια από τι μπορεί να ξεφύγει κανείς και να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας παρακαλώ λοιπόν, προτού ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε νέα μέτρα, να εξετάσουμε. Υπάρχουν τομείς όπου μπορώ να ξεφύγω με νόμιμο τρόπο και να μην βγάζει η εξάτμισή μου τελικά αυτά που απαιτεί ο νόμος. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε και νομίζω ότι το θέμα αυτό συνδέεται στενά με το θέμα της αξιοπιστίας. Ώστε να έχουμε συμμετοχή των πολιτών και να μην εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικά μέτρα στους διάφορους τομείς. Να έχουμε δηλαδή βαριά μέτρα στην ε, βιομηχανία χάλιβα ενώ να κλείνουμε τα μάτια σε άλλους τομείς. Δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα σωστά. Όσον αφορά τον επιμερισμό της προσπάθειας ε, θα υπάρξει πρόταση πριν το καλοκαίρι ή μετά. Πριν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Η Julie Γκέρλινγκ από το ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλώς ήλθατε. Θα προσπαθήσω να παραμείνω στο χρόνο ερωτήσεων. Να σας ρωτήσω πρώτα για το τσεκπομπές διοξίδιου του άνθρακος από τα Φορτίγα. Μίλησατε για τα σχέδια μείωσης της χρήσης άνθρακος και πράγματι και στο Άμστερνταμ συζητήθηκαν πολύ τα ολοκληρωμένα συστήματα για τις μεταφορές και έχουμε αυτό το τεράστιο κενό για την, ε, τον περιορισμό των ε, εκπομπών από τα φορτηγά. Ξέρω ότι για τα ελαφρά οχήματα έχετε πρόθεση να καταλήξετε σε κάτι νομοθετικά το 2017. Αυτή τη στιγμή έχουμε και θέματα ε, καταναλωτών γιατί δεν ξέρουν οι καταναλωτές αν οι εκπομπές των οχημάτων τους είναι αυτά τα οποία λέει ο κατασκευαστής και τι γίνεται με τι τοξικέ ουσίε, οι οποίε εκπέμπονται και με την οικονομία καυσίμου. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Θα πρέπει αυτή η τριπλή πρόταση λοιπόν να ε, διατυπωθεί πολύ σύντομα. Πότε μπορείτε λοιπόν να θέσετε και ενώπιον του Κοινοβουλίου την πρόταση για τις εκπομπές του άνθρωπο από τα φορτηγά και να συνοδεύονται από τα άλλα δύο θέματα που είπαμε για τα ελαφρά οχήματα και επίσης για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS για τις συζητήσεις τώρα που έχω δει να γίνονται από την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τη γαλλική πρόταση για να υπάρχει ένας κατά κάποιο τρόπο διάβλος τιμών για, το, για, τις ε, για τους ρήπους και εάν εσείς έχετε, αν σας ενδιαφέρει αυτό και αν αυτό ταιριάσει με τι προτάσει του Ηνωμένου Βασιλείου για την τιμή των καυσίμων. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τμήμα τη λύση ή είναι απλώ μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα συζήτηση που είναι ενδιαφέρουσα. Και τώρα για την ομάδα. Άλτε, ο κύριο ε, Γκέρβραντι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο για την παρουσία του για την σαφήνεια των εξηγήσεων που μας έδωσε για το τι μπορούμε να προστοκούμε από την πλευρά της Κομισιόν στον τομέα αυτό που μας ενδιαφέρει. Για τα βαρέα οχήματα είπατε ότι η Κομισιόν εξετάζει το να θεσπίσει κάποια πρότυπα για τα βαρέα οχήματα αυτό είναι, αν θέλετε, η δικιά σας, ο τρόπος να πείτε ότι θα θεσπίσετε κάποια πρότυπα. Καιρός είναι γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ιαπωνία και άλλες χώρες έχουν ήδη κάποια πρότυπα για τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Γιατί όχι και εμείς. Το κύριο ερώτημα μου όμως είναι για τη λεγόμενη φυσαλίδα άνθρακος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαν ξεκινήσει οι ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια, το έχουν αναλάβει οι κεντρικές τράπεζες, η Τράπεζα της Αγγλίας, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η δική μας τράπεζα μιλάνε για τον κίνδυνο να υπάρξει μια φυσαλίδα σε σχέση με τα θέματα του άνθρακος και η Peabody Energy στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα ε, υπέβαλε αίτηση προστασίας ε, λόγω χρεοκοπίας. Η αγορά αυτή λοιπόν έχει χάσει 97% της αξίας της μέσα σε ένα χρόνο ενώ πριν από ένα χρόνο δαπανούσε περίπου 4 ε, δαπάνησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει μια εταιρεία εξόριξης άνθρακος στην Αυστραλία. Βλέπουμε να χάνονται κάθε μέρα στην Ανατολική Ευρώπη εκατομμύρια σε, για, από εταιρείε οι οποίες ε, εξορίσουν άνθρακα. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Οι κεντρικές τράπεζες ζητούν μια ομαλή μετάβαση ε, στα ενεργειακά θέματα και όχι μια άτακτη διαδικασία που θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες της αγοράς, όπως γίνεται στην περίπτωση της εξόρυξης άνθρακος. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξή. Η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη αυτές τις εκθέσεις των κεντρικών τραπεζών. Σιάζεται μαζί με τον Ιωνάθαν Χιλ, τον συνάδελφό σας επίτροπο, να υποβάλλετε προτάσεις για να εξασφαλίσετε αυτή την ομαλή ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ. Η κυρία Στεφάνια Τόρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πράγματι με εκπλήσει που βλέπω εδώ τον κύριο Κανιέτε εδώ αυτές τις μέρες μετά το σκάνδαλο των Panama Papers όταν υπήρξαν κάποια ονόματα από την οικογένειά σας τα οποία συνδέθηκαν με αυτό το σκάνδαλο με λογαριασμούς στην Ελβετία και στον Παναμά κτλ. Εγώ θα φανταζόμουν ότι θα μπορούσατε να είχατε φανταστεί και να παραιτηθείτε. Και χαίρομαι που με βλέπετε όταν σας απευθύνω το λόγο. Θα μπορούσατε όπως έκανε ο κύριος Σόρες στην Ισπανία να ε, παραιτηθείτε. Ναι, αυτό τώρα στα ερωτήματα. Έρχομαι στο ουσιαστικό. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος στις εκθέσεις της λέει ότι η Ισπανία κάνει πολύ καλά αυτά τα οποία χρειάζονται για τον ε, μάλλον δεν κάνει τα απαραίτητα για, τον, ε, για τη μείωση των εκπομπών, αντίθετα αυξάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τι συμβαίνει λοιπόν. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσείς 80% του χρόνου σας συναντιέστε με λόμπι και όχι κανέναν άλλο και μήπως όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούνται οικονομικά οι φίλοι σας στις μεγάλες εταιρείες και όχι το να προστατεύεται η υγεία των πολιτών και ποιες εγγύησεις έχουμε επιπλέον ότι εσείς ως Επίτροπος θα διαλέξετε τα καλύτερα σχέδια υποδομών της Ισπανίας μετά από τα σκάνδαλα στην Ισπανία όπως το Ακουαμέτ που έγινε φανερό ότι το, Ευρωπαϊκό, ότι το Ποπουλάρ δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους και μετά από τα σκάνδαλα ε, τα δημοσιονομικά και διαφθοράς που έχουν να κάνουν με το Παρτίδο Ποπουλάρ στην Ισπανία, εγώ πιστεύω ότι εσείς δεν είσαστε κατάλληλος για αυτή τη θέση, το έχω πει πολλές φορές και επίσης βλέπουμε το Παρτίδο Ποπουλάρ να θεωρεί ότι τα αξιώματα είναι κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει και μια επιταγή εν λευκό. Εμείς όμως θέλουμε ο λαός της χώρας μας και όλοι οι λαοί της Ισπανίας να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να καταλάβετε πόσο μεγάλο κακό κάνετε στην Ισπανική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε για τους πρασίνους. Ζάβορ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με την χρήση της γης και με την αλλαγή της χρήσης γης που αναφέρατε στην παρουσίασή σας σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Προβλέπετε ότι δεν θα έχουμε μόνο μια αλλαγή της τάξης του 2%. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να φτάσουμε στους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, έχω θέσει το ερώτημα αυτό πολλές φορές εσάς και το θέτω και τώρα. Θα μπορούσαν να γίνουν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πιο φιλόδοξοι, να καταφέρουμε δηλαδή να μειώσουμε περισσότερο το ποσοστό αυτό και όσον αφορά την αλλαγή στη χρήση γης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει μία νομοθετική LULUCF, η οποία να συνάδει περισσότερο με το στόχο του 1,5% του 1,5 βαθμών Κελσίων συγκεκριμένα. Νομίζω λοιπόν ότι η χρήση γης, αλλαγή στη χρήση γης και τις ακομικές δραστηριότητες θα πρέπει να συνάδουν περισσότερο με το στόχο μείωσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Πολλές χώρες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο αυτό στόχο και είναι πολύ σημαντικό ο στόχος αυτό στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην, στο γενικότερο σύστημα μέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Νομίζω ότι αν αρχίσουμε να προσμετρούμε το LULUCF με τον τρόπο προβλέπεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπονομευτεί τελικά το σύστημα το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε και νομίζω ότι θα αποσταθεροποιηθεί πολύ και η όλη η αγορά εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επομένως, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένα όσον αφορά το LULUCF, Νομίζω ότι ε, ο τομέας αυτός θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος πυλώνας στο σύστημα και δεν θα πρέπει απλώς να αναμειχθεί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία προσμετρούνται. γιατί στην περίπτωση αυτή, όπως σας είπα, θα έχουμε παραποιημένα αποτελέσματα, παραπλανητικά αποτελέσματα. Για το ΙΕΝΕΦ e η κυρία Ντογνάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο διάλογος αυτός ε, είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε πώς εκτιλήσεται η συνεργασία μας και πώς αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα λοιπόν να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη οικονομική και οικολογική αλλαγή. Όλοι οι τομείς καλούνται αυτή τη στιγμή να χειρίζονται καλύτερα τους πόρους τους και να μολύνουν πολύ λιγότερο με απότερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επί της ουσίας δεν υπάρχει σημαντική απόκληση απόψεων. Το πρόβλημα έγκυται στα μέσα τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και στη μέθοδο μετασχηματισμού. Εμεί είπαμε ότι θα πρέπει να πληρώνει αυτό ο οποίο μολύνει, αυτό ο οποίο ρηπαίνει. Και επομένω το σύστημα ETS θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να μειωθεί και η διαρροή άνδρακα λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν πιο οικολογικοί οι τομεί μεταφορών και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο επιμερισμό τη προσπάθεια ανά κλάδο, ανά τομέα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Στην πράξη όμω τι βλέπουμε. Δεν υπάρχουν ε, οι απαραίτητε ε, προσαρμογές όσον αφορά τις επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν αυτή τη στιγμή από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πολύ φοβάμαι ότι ορισμένοι πολίτες και ιδίω οι γεωργοί θα καταβάλουν ένα πολύ σημαντικό τίμημα, καθότι αυξάνεται το κόστος, αυξάνονται οι δαπάνες στους ανθρώπους αυτούς και πολλές φορές πιέζονται από ένα αυξημένο ανταγωνισμό. Ιδίως ο βιομηχανικός τομέας προστιθέμενης αξίας μπορεί αυτή τη στιγμή να επηρεαστεί πάρα πολύ αρνητικά από την σκλήρινση των μέτρων ETS που προβλέπονται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει το, το πλαίσιο αξιολόγησης όσον αφορά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας αυτής και αν ε, προτίθεται να εμπλέξει περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Όλο και περισσότερο αναφερόμαστε στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Θα θέλαμε αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη και λαμβάνοντα υπόψη την υφιστάμενη οικονομική πραγματικότητα. Α είμαστε δηλαδή ρεαλιστέ και καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αναλόγω την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ. Ξαναδίνω τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις. Please express the concerns we some, some industrial sectors with the emission. Όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχουν προταθεί κάποιες τροποποίησεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά κάποιους ε, τομείς της ε, βιομηχανίας. Δαπανίσαμε πολύ χρόνο για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, μετεγκατάσταση ε, βιομηχανιών ε, εκτός Ευρώπης. Εξετάσαμε λοιπόν τους βιομηχανικούς τομείς που δαπανούν περισσότερη ενέργεια και, που, και όπου υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιοι θέλουν αυστηρή προσέγγιση, άλλοι θέλουν να προστατευτούν οι πιο εκτεθειμένοι τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή απέναντι στις προτάσεις. Θέλουμε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξετάσουμε τις οικονομικές συνέπειες οποιασδήποτε πρότασης. Διότι δεν είναι πολύ εύκολο να ταξινομήσει κανείς και να χαρτογραφήσει τις 11.000 ε, βιομηχανίες που ε, υπόγεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιον τομέα επηρεάζει τους υπολείπους. Είναι λοιπόν δύσκολη δουλειά. Γι' αυτό είχαμε ένα ολόκληρο χρόνο προετοιμασίας της πρότασης και τελικά επιλέξαμε την ε, συγκεκριμένη οδό. Πάντως ε, χαιρόμαστε το διάλογο, για το διάλογο με το Κοινοβούλιο και οι, οι, μου ε, πολύ ευχαριστώ θα εξετάσουν τον αντίκτυπο οποιαδήποτε πρόταση, Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύπλοκο νομοθέτημα αυτό. Ο κυριος ελιζε Σελίζε είπε ότι ξεχάσαμε κάποια κράτη-μέλη όταν μιλάμε για εθνικούς στόχους, Λέμε, για παράδειγμα, εντός της χώρας σας στις μεταφορές θα πρέπει να πετύχετε τον στόχο αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι μόνο σε ένα κράτος μέλος είδα περισσότερη φιλοδοξία σε σχέση από ότι ε, τα, τα επίπεδα της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει για να πετύχουμε τον στόχο αύξησης ε, της θερμοκρασίας ε, κάτω των δύο βαθμών θα πρέπει να έχουμε συνολική ευρωπαϊκή μείωση της τάξης του 30%, κάτι που θα πρέπει να γίνει με ισορροπημένο τρόπο. Σίγουρα μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε συνδέεται με τη γεωργία. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ευέλικτοι ε, που σχετίζονται με τη χρήση γης και την αλλαγή της χρήσης γης. Θα υπάρξουν λοιπόν κάποιες ε, νέες εξελίξεις όσον αφορά τους ε, μηχανισμούς ευελιξίας ε, στο πλαίσιο του Λουλουσιεφ. Όσον αφορά τις αερομεταφορές, ο Ματίας Χρότε και άλλοι είπαν ότι στο Παρίσι θέλαμε να συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές. Τελικά δεν το πετύχαμε αυτό. Θα πρέπει όμως να συμβάλλουν οι τομείς αυτοί για να πετύχουμε το στόχο της ε, αύξησης ε, της θερμοκρασίας ε, κατά λιγότερο από δύο βαθμούς. Η βάση των διαπραγματεύσεων έχει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός οδικού χάρτη. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες. που σχετίζονται ιδιαίτερα με τους στόχους ε, του 2020. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να πετύχουμε αποτέλεσμα στην ΙΚΑΟ φέτος. Και χθε είχα συζητήσεις ε, με ε, την Περιβαλλοντική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλους για να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια θέση στο πλαίσιο της ΙΚΑΟ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, σημαντικός βαθμός φιλοδοξίας από τις δύο πλευρές, ε, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της Κίνας. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την νομοθεσία να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και να προτείνει μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ε, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το χρονοδιάγραμμα μας δυσκολεύει, διότι μόλις στο τέλος της χρονιάς θα γνωρίζουμε ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην ΙΚΑΟ και αν είναι θετικό έχει καλός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών έχει δημοσιευτεί ο δικό χάρτη για να ενημερώσουμε του ενδιαφερόμενου κύκλου σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Έχουμε ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τον Μάιο και κατόπιν θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Το χρονοδιάγραμμα της πρότασης αυτής είναι πολύ σφιχτό, διότι πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της συνέλευσης του ΙΚΑΟ αρχές Οκτωβρίου και η νέα νομοθεσία θα πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2017 με τη διαδικασία της συναπόφασης. Ε, προτού προχωρήσουμε στην ε, πρώτη φάση που, στις, ε, τον Μάρτιο του 2018. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ΙΚΑΟ και θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την επίτευξη συμφωνία. Ωστόσο, κάνουμε όλη τη δουλειά που είναι απαραίτητη για να, για να υποβάλουμε τις προτάσεις μας μόλις θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στην ΕΚΑ Όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από αυτο... τα αυτοκίνητα. Και αυτό είναι ένα πολύπλοκο νομοθέτημα. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε δοκιμασίε οι οποίες δημιουργούν εμπιστοσύνη στου καταναλωτές. Η, κατα... η Κομισιόν ξέρει ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των μετρήσεων στα εργαστήρια και των μετρήσεων σε πραγματικέ συνθήκες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι αν εφαρμόσουμε την εναρμονισμένη διαδικασία για τα ελαφρά οχήματα θα αντιμετωπιστεί αυτή η απόσταση αυτό το χάσμα. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούμε να έχουμε λοιπόν πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα για τις δοκιμές αυτές, αλλά συγχρόνως η Κομισιόν εξετάζει δυνατότητα να υπάρξουν πραγματικές δοκιμασίες στο δρόμο για τις εκπομπές διοξείδιο του άνθρακος και ζητήσαμε ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις για τα θέματα αυτά από τις ομάδες εμπειρογνωμών που δημιούργησε η Κομισιόν και θα έχουμε λοιπόν τα πορίσματα προς το τέλος του χρόνου. Όταν έχουμε λοιπόν μια γνωμοδότηση για το εφικτό του να περάσουμε σε δοκιμασίες, σε πραγματικές συνθήκες, τότε θα σκεφτούμε και θα δούμε πώς μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην μελλοντική νομοθεσία για τους στόχους των εκπομπών. Ο Ματίας έθεσε ένα πολύ σωστό ερώτημα. Πότε θα έρθουν οι προτάσεις. Εμείς εργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο σκληρά για να μπορούμε να έχουμε μια πρόταση που θα έρθει σε εσά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι το μέσα Ιουλίου. Πρώτα απ' όλα θα απαιτηθεί μια μακροσκελή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, ιδίω αν έχετε και το LULUCF, την, ε, το θέμα της αλλαγής χρυσής γης. Δεύτερον, θα πρέπει εμείς να κυρώσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. 22 Απριλίου θα υπογράψουμε. Αλλά αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει αυτή τη συμφωνία, προτού τεθεί σε σε, σε εφαρμογή. Πρέπει να υπάρχουν 50 χώρες και 55% των συνολικών εκπομπών που θα κυρώσουν. Για να γίνει κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιο φιλόδοξη χώρα για τους ε, κλιματικούς στόχους και πιο ε, φιλόδοξη στην εφαρμογή, θα πρέπει να κάνει ταχαίως και την κύρωση. Αλλά βλέπουμε τώρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν ξεκινήσουν τη διαδικασία κύρωσης εάν δεν ξέρουν ήδη τους εθνικούς στόχους τους, <clears throat> γιατί αυτό θα έχει επιπτώσει στη θέση τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν καταρχήν να ακυρώσουμε τη συμφωνία και μετά να περάσουμε στους εθνικούς στόχους. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι πολλά κράτη-μέλη δεν θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ακύρωσης μέχρι να ξέρουν τους εθνικούς στόχους. Διαπραγματευόμαστε με τις χώρες αυτές και πολλοί ξέρουν ποιος θα είναι ο στόχος τους, αλλά θέλουν προηγουμένως να δούνε τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία ταχύτητος για τα φορτηγά. Κυρία Γκέρλικ, επεξεργαζόμαστε τώρα μια πρόταση για την ε, εποπτεία και, την, και τις εκθέσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι το 2017. Το 2017 θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε λοιπόν μια καλύτερη γνώση του χάσματος για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος για τα βαρέα οχήματα και θα δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε και ειδικού στόχους για τα βαρέα οχήματα. Είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση Πρώτα απ' όλα όμως θα περάσουμε στις εκθέσεις και την εποπτεία. Θα δούμε πού υπάρχουν χάσματα. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι κατά πόσο η βιομηχανία θεωρεί ότι με τόση μεγάλη, τόσο μεγάλο ανταγωνισμό στην αγορά, αν μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη απόδοση των οχημάτων. Γιατί υπάρχει ζήτηση για αποδοτικά οχήματα, αλλά παρόλα αυτά Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν συγκεκριμένους στόχους και η Κομισιόν θα πρέπει να ερευνήσει πώς οι χώρες αυτές επιτυχάνουν τους στόχους τους και πού μπορούν να βρεθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση αυτή. Μία συγκεκριμένη ερώτηση για την, τον διάβλο τιμών για τα ανώτατα όρια. Εμείς έχουμε ένα σύστημα εκπομπών το οποίο βασίζεται στην αγορά και γι' αυτό έχουμε το απόθεμα σταθερότητα τη αγορά για να μην υπάρχει πολιτική ή διοικητική παρεμβολή στην διαμόρφωση των τιμών. Θέλουμε οι τιμέ να δίνουν πραγματικά θετικά μηνύματα για τι επενδύσει σε χαμηλή χρυσή άνθρακο. Αλλά ο μηχανισμός αυτός θα έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική παρεμβολή ή επέμβαση. η Κομισιόν θέλει να έχει ένα τέτοιο σύστημα. Αν μεταρρυθμιστεί το σύστημα αυτό, θα πρέπει να γίνει και η συζήτηση στην Ευρώπη για το χαμηλότερο και το ανώτατο επίπεδο. Για ορισμένου το κατώτατο επίπεδο πρέπει να είναι και το ανώτατο επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση λοιπόν. Δεν πρέπει να γίνεται τώρα στο αυτή τη στιγμή με τα διάφορα επίπεδα. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την αρχική μας πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα στη μεταρρύθμιση του συστήματος ETS. Το Κοινοβούλιο φυσικά θα φέρει τροπολογίες. Η Κομισιόν θεωρεί ότι το απόθεμα σταθεροποίησης της αγοράς είναι ο καλύτερος δρόμος για το μέλλον και δεν θέλει να έχει οροφές και κατώ, κατόφλια. Κύριε το 2017 θα έχουμε την νομοθεσία μας για τις εκθέσεις και για την εποπτεία Χρειάστηκε πολύ καιρό η Κομισιόν να θεσπίσει αυτούς τους στόχους και τώρα θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Και τώρα αυτά που συνέβησαν με εταιρείε οι οποίε δεν ήταν μόνο εξόριξη αλλά και άλλε εταιρείε που είχαν προβλήματα πρόσφατα Α αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατάματα. Εμεί στο Παρίσι είπαμε πρέπει να περιορίσουμε την ε, αύξηση τη θερμοκρασίας σε δύο βαθμού. Αλλά ζητήσαμε και τη γνώμη του IPCC που είπε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις προσπάθειες προς το 1,5. Του ζητήσαμε να ξέρουν, να μας πούν και ποιοι είναι, ποιες είναι και οι συνέπειες του ε, να παραμείνουμε στο 1,5 1,5 βαθμούς. Το 2018 ε, θα μας κάνει και μια έκθεση για τις επιπτώσεις και μας είπαν στο Παρίσι ότι θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές μεσοπρόθεσμες για τη μείωση της, ε, της χρήσης άνθρωπος. Η Κομισιόν θα αρχίσει αμέσως μόλις έχουμε την έκθεση του 2018 του IPCC μια αξιολόγηση όλων των οικονομικών και κοινωνικών συνέπειων που θα προκύψουν από τον οδικό χάρτη της <coughs> αποανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλύσουμε όλες τις αλλαγές που θα γίνουν μέσα στην οικονομία μας για να μπορέσουμε να έχουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού με πιο καθαρές πηγές. Και αυτό έχει και συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια ενδελεχή μελέτη που θα ξεκινήσει το 2018 για να μπορούμε να στείλουμε το 2020 στα Ηνωμένα Έθνη τους στόχους μας για το μέσο του 21ου αιώνα, για όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Γι' αυτό βασιζόμαστε σε ομάδες ε, οι οποίες εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς με τον αντιπρόεδρο Κατά είναι επίσης για να δούμε και ποιοι είναι οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί αντίκτυποι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει μόνο ο Επίτροπο Ενέργεια ή Κλιματική Αλλαγή. Είναι κάτι που πρέπει να κάνει όλη η Κομισιόν με συντονισμό του αρμοδίου Επιτρόπου ω ομάδα project. Ένα πολύπλοκο εγχείρημα που θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια. Επίσης και ο Επίτροπος Χιλ θα συμμετάσχει και είναι μια μεγάλη αλλαγή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο οικονομικό σύστημα. Αν θέλετε να αποανθρακοποιήσετε την οικονομία θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, αλλά υπάρχουν συγχρόνως και μεγάλες ευκαιρίες. για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα οποία από τα Ηνωμένα Έθνη θα χρειαστούμε μέχρι το 2030 3,5-3 εκατομμύρια δολάρια επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Για τη Στεφανία Τόρες τώρα. Μου είπε, με κατηγόρησε ότι συνεργεύει πάρα πολύ με τα λόμπι. Τα εταιρικά λόμπι. Εγώ είμαι ένας επίτροπος ο οποίος δέχομαι όλους αυτούς που θέλουν να με συναντήσουμε ακολουθώντας τους κανόνες του Μητρώου Διαφάνειας και τα πρακτικά των συναντήσεων μου είναι πάντα στη διάθεση των κυρίων βουλευτών. Φυσικά, έρχομαι σε επαφή και με τη σμικιό του περιβάλλοντος, με μια τακτικότητα η οποία είναι ήδη εδρεωμένη. Σίγουρα συναντώ και αυτές τις οργανώσεις. Και φυσικά με όλους τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, ενεργειακών προϊόντων, της Ενώσης Καταναλωτών, τα συνδικάτα, με όλους αυτούς οι οποίοι μου χτυπούν την πόρτα. Αν θέλετε να δείτε πόσες συναντήσεις γίνονται στην Κομισιόν, θα δείτε ότι είμαι ένας επίτροπος με ανοιχτές πόρτες. Γιατί πρέπει να είμαι σε επαφή με την κοινωνία, με τους εμπλεκομένους, με όλους τους τομείς. Και αυτό είναι σωστό. Αν θέλετε λοιπόν να επικρίνετε δραστηριότητά μου, δικαίωμά σα να το επικρίνετε. Αν θέλετε να επικρίνετε αυτό που έκανα πέρσι, εγώ πέρσι ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο για να μπορέσω να δημιουργήσω συνένεση και να υπάρξει μια συμμαχία αυτών που, θέλουν να γίνει κάτι, που θέλουν να γίνει κάτι στο Παρίσι. Αυτό το οποίο κάνω φέτο είναι να ξεκινήσω τη διαδικασία νομοθεσίας που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους στόχους του Παρισιού σε όλους τους τομείς δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν θέλω, είναι η πρόθεσή μου να κάνω, σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι από τα πράγματα, από τα πραγματικά γεγονότα θα καταλάβετε τι γίνεται. Βλέπετε ποια είναι η νομοθεσία που θέλουμε να κάνουμε για το ETS, για την ενεργειακή μεταλλαγή, για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Είναι οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε. ο κύριος Χάμπορ. τόνισε το θέμα. Χάμπορ. Για να απαντήσω λοιπόν σε ερώτημά σα όσον αφορά τους δύο βαθμούς ή τον 1,5 βαθμό Κελσίου, επαναλαμβάνω αυτά που είπα. Θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική μέχρι το 2050 θα ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε ήδη από το 2018. Θέλουμε συνεχώς να γίνεται μία καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνουμε και των επιπτώσεων που έχουν οι αποφάσεις αυτές. Σίγουρα το Λούλουσιεφ, η χρήση της γης και η αλλαγή στη χρήση της γης, θα πρέπει και αυτό με τη σειρά του να συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ξέρετε επίση ότι και στα πλαίσια της γεωργίας είναι περιορισμένες δυνατότητε μετριασμού της κλιματική αλλαγή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό εμεί να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τη λεγόμενη περιβαλλοντική ακαιρεότητα, γιατί αν δεν ασχοληθούμε με το LULUCF, αν δεν θέσουμε ένα ανώτατο όριο, τότε μπορεί το όλο σύστημα να μην λειτουργήσει θετικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα ανώτατο όριο εκπομπών που μπορούμε να αποδεχθούμε στα πλαίσια του LULUCF. Θα υπάρχουν λοιπόν περιορισμένα επίπεδα όσον αφορά τις εκπομπές που προέρχονται από το LULUCF και από τη Γεωργία. Επίσης, αναφερθήκατε στη μείωση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα. Πάλι υποβάλλουμε μία πρόταση για το UUCF σε συνεργασία με τον Επίτροπο Χόγκαν. Τι σημαίνει αυτό. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις ανησυχίες του γεωργικού τομέα και προσπαθούμε να συντονιστούμε με τις υπηρεσίες του Επιτρόπου Χόγκαν. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση αντικτύπου και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων. Συμφωνώ μαζί σας και γενικά ως Επίτροπος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ερχόμαστε σε δημόσια διαβούλευση με τους stakeholders, με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Και θα πρέπει βέβαια να εμπλακούν και στην διαδικασία της μελέτης αντικτύπου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου, είναι αρκετά χρονοβόρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξεταστεί εκ του σύνεγγυ στη συνέχεια και επίσης ε, καταλήγουμε σε διάφορα σενάρια και διάφορες υποθέσεις προφανώς λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις απόψεις των διαφερομένων φορέων. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις αυτές, την αξιολόγηση μάλλον του αντικτύπου και να συνδυαστεί αυτό με τους πολύ φιλόδοξους στόχους που θέτουμε. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν και οι δύο αυτοί ενδιαφερόμενοι φορείς και αξιολόγηση αντικτύπου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Προτού περάσουμε στο δεύτερο γύρο μιλητών, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε 19 βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Επομένω, σας ζητώ να είστε πολύ σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Τηρήστε το χρόνο αγόρευσης. Ηβο Μπέλετ είναι ο πρώτος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Δεν θα επαναλάβω τόσο υπόθηκαν, αναφερόμενο στους τομείς που δεν υπάγονται στο ETS. Προσβλέπουμε στις προτάσεις που θα κάνετε τον Ιούλιο και υπάρχει μια έντονη διασύνδεση ανάμεσα στους κλάδους ETS και τους κλάδους που βρίσκονται εκτός ETS. Κάποια στιγμή λοιπόν το 2017 φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια κοινή απόφαση και για τις δύο κατηγορίες, έτσι δεν είναι, ETS και εκτός ETS. Αυτή τη στιγμή είδατε ότι οι περισσότεροι βουλευτέ σα ζήτησαν να είστε πιο φιλόδοξοι στον τομέα εκτό ETS, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξία όσον αφορά τον τομέα ETS. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσά να καταφέρετε να καταλήξετε πριν τι καλοκαιρινέ διακοπέ σε συμφωνία fast track με όλα τα κράτη-μέλη. Πάντω, ο κύριο Λίζ, ο κύριο Γκρότε μίλησαν για την πρόταση αυτή όσον αφορά του τομεί εκτό ETS και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε τον αεροπορικό τομέα και τις ενδοκινοτικές πτήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει στον τομέα των μεταφορών αεροπορικών, αυτιλιακών μεταφορών να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα τομέα μεταφορών πιο οικολογικό που θα περιλαμβάνει και τα βαρέα φορτηγά. Επίσης, ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι στον τομέα της ε, βιομηχανίας έχουμε εξελίξεις. Ξέρετε ότι πολύ συχνά έχουμε νέες πρωτοβουλίες βιομηχανικές οι οποίες είναι σε θέση να απορροφήσουν μεγάλα επίπεδα διοξίδιο του άνθρακα. Ας δούμε λίγο τις κοινοτόμες αυτές λύσεις. Οι καινοτόμε αυτέ λύσει αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται, δεν αποτιμούνται στα πλαίσια του ETS. Επομένω, υπάρχουν κάποιε νέε βιομηχανίε που καταφέρνουν με τι νέε μεθόδου εργασία να απορροφούν επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει και αυτέ κάπω να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό που γίνεται στα πλαίσια του ETS. Εσεί τι προβλέπετε ω προ αυτό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Παουλούτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι βασικοί στόχοι μείωση των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, εξαρτώνται πάρα πολύ από το υφιστάμενο σύστημα ETS. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι, κύριε Επίτροπε, πείτε είπατε και εσεί, συμφωνούμε μαζί σα. Παράλληλα όμω, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε με απόλυτη ειλικρίνεια ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες στρεβλωτικές επιπτώσεις στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματος ETS που είναι το βασικό όργανο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή για να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την αύξηση των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα. Αναφερθήκατε και εσεί στη διαρροή άνθρακα. Αν δούμε για παράδειγμα τον τομέα της χαλιβουργίας. Ορισμένα κράτη-μέλη έστειλαν προς τα έξω κάποιες επιχειρήσεις τους, άλλες πάλι όχι. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια στρέβλωση πάντως του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει να λεφθεί υπόψη στα πλαίσια του ETS. Σύμφωνα με την υπηρεσία anti-dumping της Ιταλίας, αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολύ ορισμένες ενωσιακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική υποστήριξη, πολλές φορές κρατική επιδότηση που λαμβάνουν ορισμένες βιομηχανίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται λοιπόν με το πρόβλημα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο, πώς καταγράφονται οι αποκλήσεις αυτές σε κοινοτικό επίπεδο, γιατί σαφώς εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην κατάρτιση των εθνικών προπολογισμών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την υφιστάμενη αυτή κατάσταση, αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενεργειακή ένωση. Ως προς αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει ένα σχετικό ψήφισμα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένους πλέον λογαριασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση που να μην επηρεάζονται από τη στρέβλωση αυτή η οποία προκύπτει αυτή τη στιγμή με το εφιστάμενο σύστημα ETS. Η κυρία Τζιψνιεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, <coughs> κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση πια. Είναι χαμηλές οι τιμές του χάλιβα που έρχονται από την ε, Κίνα και ένας από τους πολλούς λόγους για τις χαμηλές αυτές τιμές είναι η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά της Κίνας να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν μειώσεις των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος στη χώρα αυτή. Εάν η Ευρώπη θεωρήσει την Κίνα ως η οικονομία της αγοράς, τότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό των κινέζικων προϊόντων. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η άποψή σας. Ποια είναι η άποψή σας. Πρέπει να θεωρηθεί η Κίνα ως λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ποιε θα είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν για μια τέτοια απόφαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρεί η Κομισιόν ότι η Κίνα είναι δεσμευμένη να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα ακούσω βέβαια την απάντησή σας, δυστυχώς γιατί πρέπει να φύγω, θα την ακούσει ο βοηθός μου. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη για την τομέα μεταφορών. Αναφερθήκατε στις οδικές μεταφορές, αναφερθήκατε και στις αεροπορικές μεταφορές. <clears throat> Αλλά υπάρχει και το θέμα της θαλάσσιας μεταφοράς. Τι σκέφτεστε για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές και έχετε κάποια επαφή με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο, για το κλίμα παίζει μεγάλο ρόλο και η λειτουργία των ωκεανών. Υπάρχει η παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακους αλλά και η απορρόφηση από τους ωκεανούς. Το ερώτημα μου είναι, κατά τη δική σας απόψη, ποιο ρόλο θα παίξει η λειτουργία των ωκεανών για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Η κυρία Αούκεν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα. Er Δεν είναι καθόλου αυτονόητο η καύση βιομάζας να είναι βιώσιμη και ουδέτερη ως προς το διοξίδιο του άνθρακα. Υπό συνθήκες μπορεί να είναι και χειρότερο από την κάψη του άνθρακα. Βλέπουμε ότι η ζήτηση βιομάζας είναι υπερβολική και ε, πολλά κράτη-μέλη έχουν βασίσει τα σχέδια τους για αηφόρο ενέργεια στη βιομάζα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια αγορά και τον τομέα τροφίμων και μπορεί τελικά να δούμε να ε, αποψηλώνονται δάση για την παραγωγή βιομάζας. Και αυτό είναι σχεδόν το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Διότι έτσι δεν ε, θα μπορέσουμε να έχουμε απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα ε, με τους ίδιους ρυθμούς ε, που παράγεται με την καύση. Αυτό λοιπόν είναι αποφασιστική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου υποσχεθεί ότι τα κριτήρια βιωσιμότητας για την χρήση βιομάζας θα λάβει υπόψη και αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή τα έμεσα αρνητικά αποτελέσματα και όσον αφορά την απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα και όσον αφορά τη χρήση της γης. Ελπίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι θα μπορέσετε να μου υποσχεθείτε ότι θα έχουμε εξίσου αυστηρά κριτήρια για την χρήση της βιομάζας που έχουμε και για τα βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος le Κύριε Επίτροπε, στις 10 ε, Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά τις έμεσες επιπτώσεις στο έδαφος από τους υδρογονάνθρακες. Τρεις ε, επιχειρήσεις ε, παροχής συμβουλών είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Από ό,τι φαίνεται, έχει μειωθεί πάρα πολύ η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τομέα των βιοανθράκων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πάρα πολλέ θέσει απασχόληση, ιδίω στι περιοχέ τη υπαίθρου και θα μπορούσαν επίση να τονώσουν οικονομικά και κοινωνικά τι αγροτικέ περιοχέ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματεύεται μία ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες του Μερκοσούρα και προτείνει μάλιστα η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία εισαγωγή 600.000 τόνων εθανόλη σε τήσια βάση. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται εξαιτία του ILUC η παραγωγή εθανόλης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προωθούμε τελικά την εισαγωγή της ουσίας αυτής από χώρες τρίτες, τις οποίες δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος. Για ποιο λόγο δρά κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση της νομοθετικής εργασίας που προτίθεται να κάνει η Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του ETS. Εμείς θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά συγχρόνως να διατηρηθεί και η ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανιών μας και κλάδων όπως η αεροπορία όπως αναφέρθηκε. Θέλω να αναφερθώ τώρα σε μια τεχνολογία που είναι τώρα σε πειραματικό στάδιο το, η λεγόμενη power to gas, η μετατροπή της ε, ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία έχει τον ε, κάπως διακεκομένο χαρακτήρα, η παροχή ενέργειας, ιδίως από, την, ε, από τις αιωλικές γεννήτριες. πώς θα μπορούσε με την αυτή τεχνολογία να υπάρχει συσσόρευση και αποθήκευση του παραγόμενου ηλεκτρισμού από τις αιωλικές σε μεθάνιο, να μετατραπεί ο ηλεκτρισμός σε μεθάνιο που μπορεί να αποδικεύεται και να χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Η πρώτη πειραματική τέτοια μονάδα power to gas στη Γαλλία έχει γίνει στην περιοχή του mer κοντά στη Μασαλία. Τι πιστεύετε λοιπόν για αυτή την τεχνολογία που βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και αν θα ήταν έτοιμη η Κομισιόν να υποστηρίξει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καμπεθόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κανιέτε, πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όπως είπατε έχετε τον φιλόδοξο στόχο να υπάρχει ταχαίως η κύρωση της Συμφωνίας των Παρουσίων, Παρισίων και να εφαρμοστεί. Και πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα των ε, ανανεώσιμων ενεργειών, τις αποδόσεις της ενέργειας. Έχουμε όλες αυτές τις ε, προσδοκίες που έχουμε. Θα ήθελα όμως να έχω τη δική σας άποψη με ποιο τρόπο πιστεύετε θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο για την ενεργειακή απόδοση, ο οποίος θα είναι τόσο σημαντικός για το ETS. Αναφέρθηκε και εδώ το θέμα των μεταφορών για το ETS. Εδώ είναι απαραίτητο μόνο να καταμετρήσουμε τις ε, εκπομπές, αλλά να υπάρξει σημαντική μείωση των εκπομπών. Και θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει κάποια πρόταση από τη δική σας πλευρά για να, μειωθεί η, να μειωθούν οι εκπομπές από τις μεταφορές. Ένα ακόμα ερώτημα έχει να κάνει με τους καταναλωτές. Μια πρόσφατη ανακοίνωση ε, τον Δεκέμβριο του 2015 καταδείκνυε σημαντικό πως το 50% και πάνω του, τιμολογίου ηλεκτρισμού για, το μικρό, για τους μικρούς καταναλωτές είναι κυρίως φόροι των κράτων μελών. Έχουν μειωθεί οι τιμές των καυσίμων, αλλά όχι η τιμή του ηλεκτρισμού. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εσείς είχατε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια καλύτερη αντιμετώπιση και της φορολογίας της ενέργειας. Δεν ξέρω αν έχετε προχωρήσει στον τομέα αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτούς οι οποίοι πλήττονται από την ενεργειακή ένδυα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται. Υπήρξατε στο παρελθόν υπουργό Γεωργία και μιλάτε για τη σημασία τη συμπερίληψη αυτού του τομέα. Εγώ νομίζω όμω ότι εκεί πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη όχθηση προ την καινοτομία ώστε να υπάρξει και η απαραίτητη ανταγωνιστικότητα και ευελιξία για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, για την ε, παρουσίασή σας. Μιλήσατε για τη γεωργία και πράγματι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι ε, στην αλλαγή του κλίματος και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, η γεωργία μπορεί να μας δώσει τριπλό κέρδος, καταρχάς με την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και της, με τη μείωση των ε, εκπομπών, με καλύτερη χρήση των πόρων και με πιο παραγωγική γεωργία. Θα πρέπει όμως να επικεντρωθούμε περισσότερο και σε μια παραγωγή τροφίμων πιο ανθεκτική απέναντι στην αλλαγή του κλίματος ε, και να ε, επικεντρωθούμε σε καλλιέργειες ε, πιο ανθεκτικές και η γεωργία μπορεί επίσης ε, να παίξει σημαντικό ρόλο απορροφώντας τα αέρια του θερμοκηπίου. Για να το πετύχουμε αυτό όμως χρειάζεται χώρος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναπτύξουμε καλλιέργειες σε πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και με γεωργία ακριβίας μπορούμε να μειώσουμε ε, πολύ την ε, χρήση ε, των απαραίτητων πόρων. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως και πιθανές καινοτομίες για βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Θα ήθελα εσείς να μου πείτε το εξής θα δώσετε χώρο για τις καινοτομίες αυτές, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε πρακτικές λύσεις για τη γεωργία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λίνς. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ολοκλήρωση της ενεργής αγοράς ε, στην ε, Ευρώπη. Είχατε το Φεβρουάριο μία σχετική ανακοίνωση, δεν ήταν σαφές όμως εάν μιλούσατε για την δημιουργία νέων τερματικών ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποιες είναι οι δικές σας προτιμήσεις και ποιες ήταν οι αντιδράσεις από πλευράς των κρατών μελών. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι μετά την επίσκεψή σας στο Ιράν, όπου βρεθήκατε μαζί με την Υπατη ε, εκπρόσωπο, στο Ιράν ε, λοιπόν ε, υπήρξαν αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πολύ, ο Γιώλα Επίτροπε, μόλις επισκέφθηκα μια διάσκεψη για τον ρόλο των πόλεων στην προστασία του κλίματος ε, στην ε, Κίνα και υπήρξε ένα ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με τους μη κρατικούς φορείς και το ρόλο τους. Τι κάνουμε λοιπόν ε, ώστε οι πόλεις, οι περιφέρειες και άλλοι μη κρατικοί οργανισμοί να συμμετέχουν στα μέτρα για την προστασία απέναντι στην αλλαγή του κλίματος. Επίσης, όσον αφορά την βιοοικονομία. Ξέρουμε ότι γίνεται τεχνολογικός ε, αγώνας, ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην Κίνα ε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πρώτη γενιά την χάσαμε, αλλά μήπως έχουμε μια ελπίδα στη δεύτερη και τρίτη γενιά. Ίσως μπορέσει η βιοοικονομία να αποτελέσει το μέλλον μας. Εσείς τι γνώμη έχετε. Ευχαριστώ κύριο Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να ε, ακούσω την απάντησή σας. Ο βοηθός μου θα την ε, καταγράψει. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω ε, σχετικά με το κενό ανάμεσα στις πολιτικές προθέσεις μας και την πραγματικότητα. Να σας δώσω μερικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, πολλοί γνωρίζουμε ότι η χρήση του άνθρακα είναι πάρα πολύ επιβλαβής για το για το ε, περιβάλλον, ε, ωστόσο ε, βλέπουμε ότι λίγοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον άνθρακα κάτω από το έδαφος και είδαμε τώρα την πώληση από την Βάτενφαλ των εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα σε τσεχική εταιρεία, κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη χρήση. Τι θα γίνει ακριβώς αυτό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μην θέλει να τίθενται κάποια θέματα. Αυτό λοιπόν πώς συνάδει με το όραμά μας ε, όσον αφορά το περιβάλλον. Και ε, μετά έχουμε και τις μεταφορές. Ε, είναι ο μόνος τομέας όπου έχουν αυξηθεί οι εκπομπές από τη δεκαετία του 90 και ε, τελικά ε, στήριξε και το Κοινοβούλιο ε, σχετικά μέτρα. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο το κενό ανάμεσα στις πολιτικές προθέσεις μας και στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η, κυρία Ζηρικπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Επίτροπο για την παρουσία του. Ε, κάποια ερωτήματα για την ε, Γεωργία. Είπατε ότι μιλήσατε με τον ε, κύριο Χόγκαν και 40% η μείωση βασίζεται στον, στην οδηγία του 2008. Οι κάτω χώρες έχουν σημαντικές εκπομπές στον τομέα της γεωργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια γεωργία που είναι πιο φιλική από το κλίμα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη Πώς θα μπορέσει λοιπόν η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση και επικοιλία στις ανανεώσιμες ενέργειες για το βιοαέριο και την ε, βιοενέργεια. Όλα αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τη γεωργία είναι πάρα πολύ φιλικά προς το περιβάλλον και συνδέονται με την κυκλική οικονομία. Είναι σημαντικές και οι μορφές στέγασης που είναι ε, φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι βιοκλιματικές. Ε, είναι απαραίτητο όμω να υπάρξει αυτή η επιδότηση των βιοκλιματικών μορφών στέγασης, γιατί έχουμε τονίσει ότι πρέπει ο πολίτης να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να γίνει με επιδοτήσει για την ανανέωση και την ανακαίνιση αυτών των σπιτιών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζουρίνιου. Καλό απόγευμα κύριε Επίτροπε. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας για ένα ερώτημα το οποίο έθεσα χθες στον συναδελφό σας, τον κύριο Βέλο που έχει να κάνει με την πρόσφατη δημοσίευση του ενδεικτικού προγράμματος για τα πυρηνικά θέματα. Ελέγχθη ότι για την ε, τήρηση των κανόνων που είναι ενισχύ τα ευρωπαϊκά κράτη θα χρειαστούν περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025. Αυτά τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα παρά μόνο κατά το ίμιση. Η περίπτωση της Ισπανίας εδώ χρειάζονται 15 δισεκατομμύρια και μόναχα 4,3 έχουν εγγραφεί στον αντίστοιχο προπολογισμό. Είχαμε περιπτώσεις όπως το Μαράς που είχε κάποια προβλήματα ο σταθμός αυτός αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί, είναι στα σύνορα της Ισπανίας και Πορτογαλίας και οποιοδήποτε γεγονός, οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πόλεις όπως η, η Λισαβόνα. Μπορεί να υπάρξει ε, αποτέλεσμα στην ποιότητα των υδάτων, του πόσιμου υδατός. Δεν γράφουμε ποτέ στον προϋπολογισμό, δεν υπολογίζουμε ποτέ το κόστος που μπορεί να προκύψει από ατυχήματα σε αυτούς τους ποινικούς σταθμούς που εργάζονται πέραν των ορίων τους πολλές φορές και δεν χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ιβυρικής ε, Χερσονήσου. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει πιο μεγάλη ε, αποδοτικότητα αν καταλογίσουμε σωστά το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Κυρία Πιλάρ Αϊούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για το φιλόδοξο σχέδιο το οποίο μας παρουσιάζει. Έχουν γίνει σχεδόν όλες οι ερωτήσεις. Εγώ δεν θέλω να, να επαναλαμβάνω αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του χάλιβος, όπως είπαν και άλλοι. Εσείς έχετε σκεφτεί να υπάρξει κάποιος φόρος, κάποιο τέλος στα σύνορα για το εισαγόμενο ατσάλι από την ε, Κίνα και η δυνατότητα να υπάρξει κρατική βοήθεια προς τους τομείς που κινδυνεύουν από τη διαρροή άνθρακος στη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν κάποια δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αυτές οι αντικές συνέπειες. Και τέλος για τη Γεωργία αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, η Ολλανδέζα συνάδελφος, ε, μίλησε και για τον τομέα του βοήου κρέατος. Αυτά που κάνετε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Επίτροπο Χόγκαν θα λάβετε υπόψη με πού οφείλονται και σε εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες και που θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να μειωθεί το σύνολο Αυτό είναι σημαντικό θέμα, μπορεί να είναι δευτερεύον, αλλά είναι σημαντικό για τη γεωρία. Η κυρία Ντάλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Πίτο που κανιέται. Όσον αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές, αναφερθήκατε κυρίως στα βαρέα φορτηγά και απαντήσατε κυρίως στις ερωτήσεις που σας γίνουν ως προς αυτό. Να το προσεγγίσω εγώ λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Α δούμε ποιο είναι το εφιστάμενο σενάριο. Από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι και η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να είναι μια πιο βιώσιμη, οικολογική και φτηνή μορφή ενέργεια για το μέλλον, ιδίω στον τομέα των μεταφορών. Και γενικότερα συμφωνούμε ότι στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο προτίθεται να δώσει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια και πώ μπορεί να δημιουργήσει μια θετικά λειτουργούσα εσωτερική αγορά που θα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια στον τομέα των μεταφορών, γιατί αυτή τη στιγμή η φυστάμενη αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίση ότι θα πρέπει στα πλαίσια του νέου κανονισμού να χρησιμοποιηθούν και προδιαγραφέ που προέρχονται από τον Οργανισμό των Εθνών. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος, επομένως ο Επίτροπος έχει και πάλι το λόγο για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον, το ETS και τους τομείς που βρίσκονται εκτός ETS, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε πρώτα μία πρόταση για τον τομέα ETS και στη συνέχεια μία δεύτερη πρόταση για τον δεύτερο τομέα εκτός ETS. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τομέα ή αν θα πρέπει να κρατήσουμε τους δύο αυτούς τομείς ξεχωριστούς και να προβλέπετε ένα ζήτημα, ένα, ένας μηχανισμός που συγχωρείται εξισορρόπησης, αντιστάθμισης. Ξέρετε όμως ότι ε, πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται και σε αυτό το τομέα δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προφανώς και το Κοινοβούλιο αλλά και η στάση του ίδιου του Συμβουλίου. Εγώ θα προσπαθήσω σε κάθε περίπτωση να καταλήξω σε βασικές συμφωνίες επί της ουσίας και να μην φέρω από κοινού κάποιες συζητήσεις που ενδεχομένως μπορεί να περιπλέξουν περισσότερο τα πράγματα. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Καταλαβαίνω πάντως τη δική σας την προσέγγιση, όπως και καταλαβαίνω και την προσέγγιση άλλων κρατών μελών. Πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή τι αποφασίστηκε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Εγώ προσπαθώ να τηρήσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου στο δυνατόν περισσότερο. Αλλά προφανώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει αυτόνομα την απόφασή του. Επίση, στην ανακοίνωση όσον αφορά τη χαλιβουργία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συγκεκριμένη αναφορά στι νέε τεχνολογίε αποθήκευση απορρόφησης του διοξιδίου του άνθρακα. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας προς αυτό. Κάθε φορά που κάνουμε μια πρόταση και στη συγκεκριμένη αυτή πρόταση προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες επιδόσεις, ε, ποια είναι το ποσοστό χρησιμοποίησης ενέργειας ή ποιες είναι οι εμπορικές επιπτώσεις μιας ε, συγκεκριμένης βιομηχανία. Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να αντισταθμίσουμε τα πράγματα και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και τις επιμέρους αυτές ε, ομάδες, πρώτη, δεύτερη και το καθεξής, λαμβάνοντας υπόψη και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Με ορίζεται τώρα το 2020 και το Ταμείο Καινοτομίας και παντός σε όσους ε, απίφθηναν κάποιο ερώτημα όσον αφορά την καινοτομία, προφανώ θέλουμε να προωθήσουμε όλε τι καινοτόμε λύσει. Μπορούν να έχουν να κάνουν με την δέσμευση, αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα και προσπαθούμε να προωθήσουμε τις πιο τεχνολογικές λύσεις, τις οποίες υστερούμε πάρα πολλές φορές τώρα, ενώ στο παρελθόν είχαμε πολύ καλύτερες επιδόσεις. Με τον αρμόδο λοιπόν επίτροπο θα προσπαθήσω να προωθήσω περισσότερο τις καινοτόμε τεχνολογικέ λύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, στον τομέα της χαλιβουργίας υφίσταται ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα. Και ο πιο καθοριστικός παράγοντας, θα έλεγα, δεν είναι τόσο πολύ τιμή του άνθρακα στα πλαίσια του κανονισμού ETS. Στο παρελθόν, άλλωστε, είχαμε πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων εκπομπών και το πρόβλημα τώρα είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή Έχουμε μια πλεονάζουσα παραγωγή από την Κίνα που επηρεάζει προφανώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή φανιζόμαστε εμείς να είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα αυτό. Θέλουμε επίσης να δούμε και το νέο σχεδιασμό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την νέα νομοθεσία θα έχουμε μια πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας με χαμηλότερες τιμές και υψηλότερο ανταγωνισμό. Όσον αφορά τώρα Ένα άλλο ερώτημα που μετέθη όσον αφορά το καθεστώ οικονομία τη αγορά τη Κίνα, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει όλε τι επιπτώσει που θα έχουμε από την ε, αναγνώριση ενό τέτοιου καθεστώτο αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως ξέρετε, για την χαλιβουργία και αργότερα θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα των επιπτώσεων εφόσον να γνωριστεί το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Η κυρία Μέσνερ στη συνέχεια έκανε ένα ερώτημα για τις μεταφορές και όντως δεν κάλυψε επαρκώς το ναυτιλιακό τομέα. Δεν αναφέρθηκα σε αυτόν. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός προσπαθεί και αυτός να έχει πιο συγκεκριμένου κανόνες παρακολούθησης των θαλασσίων μεταφορών. Πρέπει λοιπόν και με τον οργανισμό αυτό, όπως και με τον ΙΚΑΟ, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε ένα μνημόνιο συνεννόησης. Γιατί ξέρετε ότι ε, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και με τον ΙΚΑΟ και με τον IMO. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία του Παρισιού. Συντονιζόμαστε επίσης προφανώς και με τον Επίτροπο Βέλα και για το ζήτημα αυτό. Η κυρία Άουκιν στη συνέχεια έθεσε ένα ερώτημα όσον αφορά τη βιομάζα, αν δεν κάνω λάθος. Μα βεβαίως, βεβαίως, η βιομάζα μπορεί να τραυματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και Ξέρω ότι ε, στα πλαίσια της ε, οδηγίας για την βιομάζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε κάποια ζητήματα με ορισμένα κράτη-μέλη. Συνεργάζομαι και με τον Επίτροπο Χόγκαν και με τον Επίτροπο Βέλα και στα πλαίσια της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμπεριλάβουμε και τη βιομάζα μέχρι τα τέλη του 2016. Προφανώς θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τα ασφάλματα του παρελθόντος. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη που είχαμε κάνει και στα πλαίσια του ILUC, όπου δώσαμε κάποια λανθασμένα, λανθασμένες ενδείξεις όσον αφορά τι επενδύσει και χρειάστηκε στη συνέχεια να υπαναχωρήσουμε στις ε, αρχικές μας θέσεις. Η βιομάζα πάντως θα πρέπει να αποτελέσει μελλοντική πηγή ενέργειας, αρκεί βέβαια να είναι βιώσιμη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντική ακαιρεότητα και βιωσιμότητα της βιομάζας. Περνάω σε ένα ακόλουθο ερώτημα το οποίο είχε να κάνει με το ILUC. Απάντησα πάνω στο ερώτημα αυτό, αναφέρθηκα και στο φυσικό αέριο. Προφανώς θέλουμε να προωθήσουμε κάθε μορφή καινοτομία, η οποία θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τις ικανότητες αποθήκευσης είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε όσο δυνατόν υψηλότερες ικανότητες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα και αυτό να συνδυάζεται με τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βέβαια αυτό συνδυάζεται και με την παραγωγή φυσικού αερίου για το μέλλον. Η κυρία... Η κυρία Καμπεθών τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των μεταφορών. Εμείς θα εκδώσουμε και μία ε, ανακοίνωση για τη μείωση της χρήσης άνθρακος στον τομέα των μεταφορών για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης μέσα στα πλαίσια των εφιών συστημάτων των αυτομάτων αυτονόμων και εφιών συστημάτων μεταφορών για όλες τις υποδομές οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά το κλειδί είναι η καινοτομία. Να έχουμε την πιο αποτελεσματική χρήση μέσω μεταφοράς όχι μόνο στα οχήματα, αλλά για, γενικά για τη διαχείριση των ροών των μεταφερικών ε, ε, φορέων. Να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας. Πολλοί βουλευτές μίλησαν για το θέμα αυτό. Μίλησαν πολύ λοιπόν για την ηλεκτροκίνηση και εδώ είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι να αντιμετωπίσουμε ότι είναι πιο ακριβά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν υπάρχει αρκετή υποδομή για τη φόρτιση των οχημάτων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, δυσκολία και ένα από τα θέματα είναι να μας ε, να αντιμετωπίσουμε και στα πλαίσια της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων όλα τα νέα κτίρια να έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν αυτοκίνητα. Παραδείγματος χάρη το, το γκαράζ των οχημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πόσες θέσεις υπάρχουν για φόρτιση και πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, σε άλλους τομείς θα πρέπει εκεί πέρα να δημιουργήσουμε την υποδομή για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και στους αυτοκινητοδρόμου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία να υπάρχουν τέτοια σημεία φόρτιση στους αυτοκινητοδρόμου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Πρέπει να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Και σίγουρα υπήρξε το ερώτημα του κ. Λίμπερ για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Εκεί η Κομισιόν αυτό το οποίο προσπαθεί είναι να έχει ασφάλεια εφοδιασμού. Χρειαζόμαστε πιο πολύμορφους ε, δρόμους εφοδιασμού και πάροχους. Έχουμε μια στατηγική για το φυσικό αέριο ως Κομισιόν που έχουμε διατυπώσει και θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες διασυνδέσεις να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό το οποίο είναι στη διάθεσή μας και να έχουμε και περισσότερες διασυνδέσεις ώστε να έχουμε ένα γενικό σχέδιο για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Όταν πήγα στο Ιράν πήρα το μήνυμα ότι θέλουν να ε, έχουν εξαγωγές ε, αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι πολύ δύσκολες οι ε, διαπραγματεύσεις με τις χώρες διέλευσης των αγωγών φυσικού αερίου και θεωρούν ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορες εξαγωγές γιατί θα δημιουργηθούν τρία τέτοια κέντρα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είχαν σταματήσει ήδη από την εποχή της Ιρανικής Επανάστασης αλλά τώρα μπορούν να προχωρήσουν. Ο κ. Λέιντεν αναφέρθηκε για τις οικονομίες στα καύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έχουμε τον οριζοντά 2020 όπου τονίζουμε την καινοτομία αλλά έχουμε και τα συστήματα ρύθμισης τα οποία πρέπει να λυθούν. υπόψη. Θέλουμε οι φορείς να έχουν ένα σταθερό ρυθμιστικό οριζόντα ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν. Ο κύριος ε, Σελίμοβιτς μίλησε για το Nord Stream 2. Δεν ακολουθεί απόλυτα τους στόχους ε, διαφοροποίησης για, τους, ε, για την παροχή φυσικού αερίου που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το να έχει τα 80% της παροχής φυσικού αερίου από την ε, Ρωσία, είναι αντίθετο με αυτούς τους στόχους. Θέλουμε να έχουμε και διέλευση και από άλλες περιοχές όπως η Ουκρανία. Νομίζουμε ότι όλη η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αφορά στις δημόσιες προμήθειες είτε αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά για τον αγωγό αυτό. Ο κ. Ζουρίνιο αναφέρθηκε στους πυρηνικούς σταθμούς, μα η έκθεση αυτή για τους πυρηνικούς σταθμούς είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν να κάνει μια έκθεση και δεν είναι πολιτική αξιολόγηση, λέμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση αλλά η ασφάλεια των ποινικών σταθμών είναι η ευθύνη των κρατών μελών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και η Κομισιόν έχει τρεις οδηγίες για τα θέματα. Έχουμε τονίσει ιδιαίτερα τα θέματα αυτά μετά την Φουκουσίμα. Αλλά είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν στα θέματα αυτά. Και η Κομισιόν παρακολουθεί όχι μόνο αυτό τον ποινικό σταθμό, αλλά και άλλους στο Λουξεμβούργο ή στις βαλτικές χώρες. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και εμεί θέλουμε να έχουμε το πιο φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο και ζητούμε από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να το εφαρμόσουμε. Στην κυρία Πιλάρα Ιούσο, κάνετε το πιο δύσκολο ερώτημα. αναγνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά και τα επεξεργαζόμαστε και τέλος τι είπε η κυρία Ντέιλι δεν μπορώ να διαβάσω και τα γράμματά μου μιλήσατε για τον ηλεκτρισμό και μιλήσατε και για τη φορολογία αυτό το οποίο θα κάνει η Κομισιόν για τον ηλεκτρισμό και το τίμημα του ηλεκτρισμού Θέλουμε να έχουμε μια αγορά χωρίς προσκόμματα. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια επαρκή δυνατότητα παραγωγή όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει ένα μηχανισμό υποστήριξη, ίσω όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η τιμή του ηλεκτρισμού έχει σχέση με το κόστος. Όπως είπε και η κυρία Καμπεθόν, θα πρέπει, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ενεργειακής ένδειας. Ο αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς είναι πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας με πολλούς πολλούς επιτρόπους που αναλύουν πώς θα καθορίσουμε την έννοια της ενεργειακής ένδειας με εναρμονισμένο τρόπο και πώς θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά της ενεργειακής ένδυας. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπόρεσα να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις αλλά ίσως κάποια ερωτήματα έχουν μείνει ανοιχτά και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να απαντήσουμε για τα προβλήματα του μεθανίου στην Γεωργία. Φυσικά όταν υπολογίζουμε την ε, επίπτωση της αλλαγής υγιής και την αποψήλωση λαμβάνουμε αυτό υπόψη και λαμβάνουμε υπόψη τη δυνατότητα να μειώσουμε με, ε, σε άλλους τομείς για να αντισταθμίσουμε την αύξηση των εκπομπών στη γεωργία. Θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά και με την καινοτομία μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά και εμείς υποστηρίζουμε κάθε μορφή καινοτομία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις σας, για την παρουσία σας εδώ και για τις προσπάθειες που καταλάβατε, καταβάλατε να απαντήσετε στον δω περισσότερες από τις ερωτήσεις. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Και ευχαριστούμε και πάλι τον Επίτροπο για την παρουσία του και τονίζω και πάλι τη σημασία του διαφρομένου διαλόγου. Θα τα πούμε το απόγευμα.